πάμε αμέσως στην πιθανή επιβολή θανατικής ποινής στον Ιμπραήμ Χαλάουα. Το λόγο έχουν οι συντάκτες. Πρώτος, για ένα λεπτό, ο κύριος Κοράου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο Ιμπραήμ Χαλάουα Ξέρετε ότι κατα... κατηγορείται και ενδέχεται να του επιβληθεί η θανατική ποινή επειδή συμμετείχε σε μία διαμαρτυρία. Ας μιλήσουμε σαφώς από τότε που αλσίζει κυβερνά την Ευρώπη, ξέρουμε ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να προωθήσουμε έναν καρποφόρο διάλογο με τη χώρα και λόγω γεωστρατηγικής θέσης, αλλά δεν μπορούμε να δεχτούμε να χρησιμοποιούνται τέτοιοι νόμοι επιβάλλοντας θανατική ποινή για σήμαντους λόγους Ξέρουμε ότι πολλά κράτη-μέλη ε, έχουν ξεκινήσει ένα διάλογο με την Αίγυπτο έτσι ώστε ο Ιμπραήμ να απελευθερωθεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει για ένα λεπτό ο κύριος Ντέμες Μάκερ. Συνάδελφοι, σε ένα κελί στην Αίγυπτο, βασανισμένος, χτυπημένος. Ε, έτσι πέρασε λοιπόν ο Ιρλανδός υπήκος Ιμπραήμ Αλάβα τα γενέθλιά του. Και γιατί, γιατί χρησιμοποίησε το δικαίωμά του για ελευθερία ε, έκφρασης, ε, ελευθερία συνάθρησης και με την απεργία πείνας τώρα λοιπόν ζητά την ε, προσοχή της διεθνούς κοινότητας. Οι εκλογές του 2011 ήταν για πρώτη φορά ε, φωνή σε εκατομμύρια ανθρώπους. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι αδερφοί μουσουλμάνοι δεν άκουγαν τους αντιφρονούντες, αλλά τα πηγαίνει καλύτερα άρα για το σημερινό καθεστώς. Είναι λιγότερο αυτοκρατικό, λιγότερο καταπιαστικό. Οι προσωπικές ελευθερίες και οι ελευθερίες του πολίτη είναι ακόμα πιο περιορισμένες σήμερα από ότι υπό το Μουμπάρακ. Η απειλή της αντικής πυλής ξεπερνάει οποιαδήποτε όρια δεν συνάδει με την πλειοψηφία αυτό που ζητούν οι Αιγύπτιοι. Ένα σταθερό και ελεύθερο δημοκρατικό καθεστώς. Καλό λοιπόν τις Αιγυπτιακές αρχές να δώσουν μια δίκαιη δίκαιη στον Χαλάβο και στους 400 άλλους στους κρατουμένους. λεπτό η κυρία Σαρτζεντίνη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο Ιμπραήμ Χαλάβα συνελήφθη όταν ήταν 17. Πρόκειται για ένα παιδί. Υπάρχουν διεθνείς κανόνες για το πώς αντιμετωπίζει κανείς τα παιδιά στις φυλακές. Πώς τα μεταχειρίζεται. Έχουν περάσει κάποια χρόνια έκτοτε και δεν τα πηγαίνουν καλά. Ούτε οι άλλοι εκατοντάδες αληφθεί και βρίσκονται στις φυλακές, οι οποίοι δεν ε, περνούν από μαζικές δίκες και δεν ε, ξέρουν καν τι γίνεται με τις υποθέσεις τους και τι κατηγορίες τους απαγγέλλονται. Αυτή είναι λοιπόν η σημερινή Αιγυπτός και αυτή είναι η Αιγυπτός για την οποία πολλοί συνάδελφοι λένε ότι θα πρέπει να συνάψουμε συμφωνίες. Η Αίγυπτος με την οποία θεωρούμε ότι είναι στρατηγικός τέρος μας σε μια ασταθή περιφέρεια που θα μας βοηθήσει να σταθεροποιήσουμε την περιφέρεια. Μα είναι τραγικό το λάθος αυτό. Πρόκειται για μια χώρα που απεσταθεροποιεί και ε, ο είναι ο Μουμπάρακ υπαριθμών 2 ο κόσμος αγανάκτησε και μετά από δεκαετίες καταπίεσης εξεγέρθη κατά του Μουμπάρακ και θα αναγκαστεί να το ξανακάνει. Και εμείς αποστρέφουμε το βλέμμα μας. Ελπίζουμε να απελευθερωθεί ο Ιμπραήμ Χαλάβα, αλλά αποστρέφουμε το βλέμμα μας από αυτά που συμβαίνουν ε, στο, στην Αιγυπτό. Νέτσετς Σιτόρτον και Ντόμινικ Κέιν. Ευρωπαίοι δημοσιογράφοι που καταδικάστηκαν χωρίς ε, δίκη. δίκη. Και αυτοί λοιπόν αξίζουν ε, τη δικαιοσύνη. Το λόγο έχει για ένα λεπτό η κυρία Χάρκη. Ευχαριστώ. Ε, έχω πολλά κοινά με τον Ιμπραχήμ Χαλάουα. Και οι δύο είμαστε Ιρλανδοί. Και οι δύο είμαστε Ευρωπαίοι πίκοοι. Και στο πλαίσιο αυτό και κυρίως επειδή ο Ιμπραήμ Χαλάου ήταν ανήλικος όταν συνελήφθη, ζήτησε από τις Αιγυπτιακές Αρχές ε, άμεσα και ανεφόρον να αποφυλακίσουν τον ε, Ιμπραήμ Χαλάουα και χρησιμοποίησε τους όρους πάραφτα και ανεφόρων γιατί έχει μείνει μέχρι στιγμής 849 ημέρες στη φυλακή και 10 φορές έχει αναβληθεί δίκη του και μάλιστα χρησιμοποίησε τους όρους ε, πάραφτα και ανεφόρων γιατί ε, ο Ιμπραήμ Χαλάου ακρίθηκε ως φυλακισμένος ε, για ιδεολογικούς λόγους από τη Διεθνή Αμνηστία. Μάλιστα θα, ε, θα δικαστεί από κοινού με 493 άλλους ανθρώπους χωρίς καμία εγγύηση για δίκαιη και ελεύθερη δίκη. Χρησιμοποίησε λοιπόν τους όρους πάρα και ανεφόρων γιατί η Ιρλανδική κυβέρνηση ζήτησε την αποφυλάκησή του με το Προεδρικό Διάταγμα 140. Ζητώ λοιπόν ενίσχυση των προξενικών ε, διαβημάτων από τις Ιρλανδικές Αρχές. Και ευχαριστώ τους συναδέλφους που έθεσαν το θέμα πολλές φορές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ευχαριστώ και τον Γκλιμ ε, Μπόιλον ε, που φρόντισε ώστε το όνομά του και η υπόθεση Χαλάουα να μην διαφύγει της προσοχής μας. Ευχαριστώ. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω όλες τις πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη συνεργασία τους στην εκπόνηση ε, του ψηφίσματος που συντάχθηκε με ομοφωνία. Επίσης να ευχαριστήσω τους συνεισηγητές, κυρίως ε, τη Μάριαν Χάρκιν και, τον, ε, και την Λίν Μπόιλαν. Και ευχαριστώ γιατί μας βοήθησε και η οικογένεια του ενδιαφερομένου να ε, συντάξουμε το ψήφισμα και να επιστήσουμε την προσοχή μας σε αυτή την περίπτωση. Η περίπτωση του Ιμπραχήμ Χαλάουα είναι απολύτω απαράδεκτη. Ένα 17χρονο ανήλικο Ιρλανδό υπήκο συνελήφθη στι διαδηλώσει στο Κάιρο το 2013, συνελήφθη και έκτοτε παραμένει στις φυλακές σε άθλιες συνθήκες. Κάτι τέτοιο αντιβαίνει στο, στην διακήρυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα των ανηλίκων. Και ε, η Ιρλανδική κυβέρνηση και ο Υπουργό Εξωτερικών τη Ιρλανδία προσπάθησαν να πείσουν τι Αιγυπτιακέ Αρχέ ε, να επιλύσουν το ζήτημα αυτό το συντομότερο δυνατόν, ώστε να επιστρέψει ο Ιμπραήμ Χαλάουα στην πατρίδα του την Ιρλανδία. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει για ένα λεπτό η κυρία Λίν Um, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να καλωσορίσω καταρχάς ε, την αδερφή του Ιμπραχήμ Σομάγια που ήλθαν να, να εκπροσωπήσουν τον αδερφό τους και με τους οποίους συνεργαστήκαμε τα δύο χρόνια. Το ψήφισμα αυτό καταδικάζει δικαίως το γεγονός ότι ο Μπρεχήμ ανήλικος όταν συνελήφθη αντιμετωπίζει μια μαζική δίκαια στην οποία ούτε μόνο, όχι μόνο δεν μπορεί να ματρήσει αλλά ούτε να συμμετάσχει και να ακούσει την ε, δίκη. Και καλώς ορίζω το γεγονός ότι όλες οι πολιτικές ομάδες και ιδιαίτερως όλοι οι Ιρλανδοί συμφωνούν Έχουμε συζητήσει το περιεχόμενο της υπόθεσης του Ιμπραχήμ θα ήθελα λοιπόν να αναφέρω το τι μας ε, μετέφερε μυστικά ο Ιμπραχήμ ε, από τη φυλακή. Για τρίτη φορά λέει βρίσκομαι στα γνέθλιά μου στη φυλακή και θα ήθελα να δώσω τις ευχές μου στην, ε, με την ευκαιρία αυτή προς όλους όσους υπερασπίζονται τις ανθρώπινες ελευθερίες που ανάβουν ένα κερί κάθε βράδυ για να θυμούμαστε ότι δεν μπορούμε να καταπιεστούμε κάθε βράδυ προσεύχομαι και πρέπει οι τεκεριά αυτά να φωτίσουν το μονοπάτι της ελευθερίας. Σας ευχαριστώ κυρία Μπόιλαν. Το λόγο έχει για ένα λεπτό επίσης ο κύριος Παντσέρη. Ευχαριστώ. Ο Ιμπραήμ Λάουα έχει να αντιμετωπίσει μία πολύ δύσκολη δίκη και το ενδεχόμενο της θανατικής ποινής, γιατί τον Αύγουστο του 2013 συμμετείχε σε μία διαδήλωση στο Κάιρο. Τότε ήταν 17 χρονών, άρα ανήλικος. Παρ' όλα αυτά, το Αιγυπτιακό Δικαστήριο δεν το δέχτηκε υπόψη, παραβιάζοντας την Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Παιδιών. Ξέρουμε ότι βασανίστηκε κατά την κράτησή του και κρίθηκε ένοχος. Το Μάιο του 2015 καταδικάστηκαν σε θανατική ποινή πέντε άνθρωποι οι οποίοι έχουν την ίδια ηλικία με τον Ιμπραήμ. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τη στιγμή της υποτίθεται αξιόπινης πράξης ήταν 17 χρονών. Είμαστε πολύ ανήσυχοι και ζητάμε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 όλους για τη μάχη που δίνουν εδώ και ε, χρόνια και ιδιαίτερα της κυρίας Μπόιλεν. Δεν πρόκειται μόνο για έναν Ιρλανδό πολίτη όπως είπε η κυρία Χάρκιν. Είναι και Ευρωπαίος. Η Ευρώπη βασίζεται στην ελευθερία, δικαιώματα και αναφέρετα ανθρώπινα δικαιώματα που εγγράφονται στο ευρωπαϊκό δίκαιο. Θεωρούμε λοιπόν ότι θα πρέπει και οι τρίτες χώρες με τις οποίες έχουμε σχέσεις να υπερασπιστούν αυτά τα δικαιώματα. Θα ήθελα να λάβουν υπόψη οι Αιγυπτιακές αρχές ότι το Κοινοβούλιο μιλάει με μία φωνή σήμερα και θα ήθελα να χρησιμοποιήσουν το νόμο 140 με βάση τον οποίο με ένα προεδρικό διάταγμα ο, Ιμπραχα, ο Ιμπραήμ Χαλάουι θα μπορούσε να έρθει στη χώρα του σήμερα και να απελευθερωθεί άμεσα. Θα ήθελα να ρηχτεί φως σε αυτή την υπόθεση. Σοσιαλιστών και Δημοκρατών έχει ο κύριος Βάιντεν Χόλτζερ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο Ιμπραχήμ Χαλάβα αποτελεί μια τραγική υπόθεση γιατί τα καταδεικνύει τι μπορεί να συμβεί σε ένα άτομο όταν τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου δεν ε, τηρείται και οι Αιγυπτιακές αρχές ε, θα πρέπει σε αυτή την περίπτωση αυτή να αποδείξουν το αντίθετο. Ο Ιμπραχήμ Χαλάβα ωστόσο δεν είναι μια μεμονωμένη υπόθεση. Υπάρχει μια συστηματική καταπάτηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των αρχών του κράτου δικαίου στην Αίγυπτο και αυτό μα πονάει ιδιαίτερα γιατί συμβαίνει στην Αίγυπτο, γιατί η Αίγυπτος είναι σημαντικός εταίρο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί εκτιμούμε τι ε, προσπάθειε κατά τη τρομοκρατία που γίνονται από την Αίγυπτο και γιατί θέλουμε να υπάρχει σταθερότητα στην Αίγυπτο, αλλά η πραγματική σταθερότητα, αγαπητοί συνάδελφοι, μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν τηρείται η δημοκρατία. Η Ιτάλος ε, η χύτρα ταχύτητος κάποια στιγμή θα εκραγεί. Για την ομάδα των φιλελευθέρων και δημοκρατών το λόγο έχει για ένα λεπτό η κυρία Σκάκη. Ευχαριστώ Πρόεδρε, συνάδελφοι, Επίτροπε. Στην Αίγυπτο τα βασικά δικαιώματα, η δίκαιη δίκη είναι δικαιώματα τα οποία καταπατώνται και το καθεστώς έχει προκαλέσει πάρα πολλά θύματα. Στην Αίγυπτο οι ακτιβιστές μας λένε ότι τα πράγματα είναι χειρότερα από ό,τι ήταν ε, υπό τον πρόεδρο Μουμπάρα και δεν θα πρέπει να αποστρέφει το βλέμμα της η Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί αυτό δεν είναι μια λανθασμένη αίσθηση σταθερότητας η οποία δεν είναι βιώσιμα. Η μουσουλμανική αδερφότητα προωθεί ε, την, ε, τον πλουραλισμό, τη δημοκρατία. Όχι, δεν το πιστεύω αυτό. Με ανησυχούν οι πολιτικές των κινημάτων αυτών. Ωστόσο, θα έπρεπε να θεωρείται αθώος μέχρι αποδείξεως τον, εναντί, του, αντιθέτου ο Χαλάβα Και σε μαζικές δίκες δεν μπορεί να υπάρξει πραγματική δικαιοσύνη. 420 άτομα θα εκδικαστούν την, ε, ε, εκδικάστηκαν μάλλον την ε, Κυριακή και αναβλήθηκαν λοιπόν οι δίκες αυτές επειδή δεν ήταν παρόντες. 17 λοιπόν ήταν ο κύριος Χαλάουα όταν συνελήφθη. Και γι' αυτό λοιπόν ζητούμε να απελευθερωθεί βάση του διατάγματος 140. Ελευθερίας και άμεσης δημοκρατίας για ένα λεπτό η κυρία Τζέιμς. Good morning. Καλημέρα σας. Οι Βρετανοί Μιλάνε για τον ελέφαντα που βρίσκεται μέσα στην αίθουσα, ενώντας ότι κάτι είναι οφθαλμοφανές, αλλά κανένας δεν το λαμβάνει υπόψη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει το δικό της ελέφαντα στην αίθουσα και είναι η Τουρκία. Και το τονίζω αυτό γιατί κάθε φορά μιλάμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Στρασβούργο. Σήμερα μιλάμε για τον κύριο Χαλάουα. Όμως η Τουρκία είναι η χώρα που έλαβε τρία ε, δις ευρώ για να αντιμετωπίσει το προσφυγικό, αλλά δεν μπορεί να τηρήσει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα ήθελα κάτι να βγει το θετικό από τις ομιλίες σήμερα το πρωί, αλλά νομίζω ότι μιλάμε για δύο μέτρα και δύο σταθμά αν επιλύσουμε, μόνο αν επιλύσουμε το ζήτημα που ετέθη σε σχέση με την προσχώρηση της Τουρκίας, δεν θα επιλύσουμε το θέμα των διπλών μέτρων και σταθμών που ισχύουν για την περίπτωση Χαλάουα και άλλων που παραβιάζουν ανθρώπινα δικαιώματα. Το λόγο έχει για 1,5 λεπτό ο κύριος Επιτίδιος, μία εγγεγραμμένος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε ο Ιμπραήμ Χαλάουα είναι νεαρό νεαρός Ιρλανδοαιγύπτιος, ο οποίο κρατείται από το 2013 σε φυλακή του Καΐρου μαζί με άλλα 492, 93 άτομα, κατηγορούμενο για σωρία ποινικών αδικημάτων που περιλαμβάνουν καταστροφή και φθορά δημοσία περιουσία, ακόμη και δροφωνίε πολιτών. Σύμφωνα με τα στοιχεία τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω έχουν παραβιαστεί τα ανθρώπινα δικαιώματα του κυρίου Χαλάουα, διότι αυτό κρατείται επί δύο χρόνια χωρί ακόμη να έχει καθοριστεί η δίκη του, έχει υποστεί βασανιστήρια το έχει στερηθεί η δυνατότητα ιατροφαρμακευτικής περιθάλψεως και τέλος αντιμετωπίζει τον κίνδυνο ε, του θανάτου αν και όταν συνελήφθη ήταν 17 ετών μόλις. από την πλευρά της η αίγυπτος αναφέρει ότι δεν έχουν παραβιαστεί τα ανθρώπινα δικαιώματα του κυρίου χαλάουα αναφέρει τα ε, αδικήματα τα οποία έχει υποπέσει αφήνει να νοηθεί ότι θα τύχει δίκαια δίκη και ενδεχομένω ο πρόεδρο τη δημοκρατία να τον απαλλάξει από την έκτηση του υπολείπου τη ποινή όταν ανακοινωθεί το αποτέλεσμα τη δίκη. η υπόθεση χαλάουα είναι μία από τι πολλέ περιπτώσει παραβιάσεω των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλο τον κόσμο. η άποψή μου είναι ότι η ευαισθητοποίηση και η κινητοποίηση τη ευρωπαϊκή ενώσεω σε συνδυασμό με το γεγονό ότι την υπόθεση Χαλάου την παρακολουθούν στενά οι υπάλληλοι του προξενιού ε, της ιρλανδίας στο κάιρο θα έχει ως αποτέλεσμα την απελευθέρωση του κυρίου Χαλάου ασχέτως του αποτελέσματος της δίκης. άλλωστε η αίγυπτος είναι μια από τις χώρες που έχει στενές οικονομικές και πολιτικές σχέσεις με την ευρωπαϊκή ένωση και δεν θα θελήσει να τις ε, ε, καταστρέψει χάρη του κυρίου Χαλάου. Εκείνο που πρέπει να μας ενδιαφέρει είναι να βρούμε και να θεραπεύσουμε και να δικαιώσουμε πολλέ περιπτώσει ανθρώπων που μοιάζουν με, την, ε, με τον κύριο Χαλάου αλλά δεν είναι ακόμη γνωστοί. Τέλο, καλό θα είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση να φροντίσει να μην παραβιάζονται τα δικαιώματα των ε, Ευρωπαίων πολιτών στα κράτη-μέλη τη, κάτι το οποίο όπω γνωρίζετε πολύ σωστά, ε, πολύ καλά έχει συμβεί στην πατρίδα μα με θύμα το δικό μα κόμμα. Σα ευχαριστώ. το λόγο έχει για ένα λεπτό ο κύριο Βέντα. Ευχαριστώ. Ο Ιμπραήμ Χαλάουα ήταν 17 ετών όταν συνελήφθη και υπέστη επίθεση και από τις ε, δυνάμεις ασφαλείας. Τον απειλεί θανατική ποινή. Και μάλιστα τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί η εκτέλεση των θανατικών ποινών. 12 άτομα έχουν φέτος εκτελεστεί. Ουσιαστικά καταστρατηγήθηκαν τα δικαιώματα ελεύθερης έκφρασης, το δικαίωμα του συναθρίζεστε, από τις Αιγυπτιακές αρχές. Ο Ιμπραήμ Χαλάουα ξεκίνησε και απεργία πείνας. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει ε, δίκαιη και ελεύθερη δίκη με βάση τις ε, διεθνείς προδιαγραφές. Επίσης ε, υπάρχουν πολλές υπόνοιες ότι πέστη και βασανιστήρια ο κύριος Χαλάουα. Είναι κατάφορη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ενός Ευρωπαίου πολίτη. παραβιάζεται μάλιστα και η Διεθνή Σύμβαση για την απαγόρευση τη εφαρμογή βασανιστήριων και απάνθρωπων και ξεφτυλιστικών συμπεριφορών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η περίπτωση καταστρατήγηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αίγυπτο δημιουργεί φοβερέ ανησυχίε. Οι Αιγυπτιακέ αρχέ ε, περιφρονούν ουσιαστικά ανθρώπινα δικαιώματα, όπω είναι η ελευθερία του συναθρίζεσαι, η ελευθερία έκφραση. Και μάλιστα ένα ανηλίκος εδώ και δύο χρόνια είναι φυλακισμένος χωρίς να το έχει απαγγελθεί κατηγορία, ενώ, ε, χωρίς να το έχει γίνει δίκη, ενώ τον απειλεί και θανατική καταδίκη. Ε, νομίζω ότι θα πρέπει ε, να ε, επισημάνω αυτή την ε, κατάφορη καταστρατήγηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μάλιστα τον ε, Αύγουστο του 2013 οι αρχές της ασφάλειας αφάρμοσαν βία κατά ειρηνικών δηλωτών με πολλούς νεκρούς και πάρα πολλούς τραυματίες. Ε, καταπατείται λοιπόν κατάφορα η ελευθερία έκφρασης και η ελευθερία συνάρτησης. Συζητούμε από την Αίγυπτο να αποφυλακίσουν πάραυτα όλους τους πολιτικούς ε, κρατουμένους. Γιατί με βάση την Διεθνή Διακήρυξη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα σε ελεύθερη, δημόσια και ε, δίκαιη δίκη από αμερόληπτο δικαστή. Θα πρέπει και η Αίγυπτος να τηρήσει αυτές τις αρχές. η σειρά των εγγεγραμμένων Έχω δεχθεί τρία αιτήματα με τη διαδικασία του Catch the Eye. Επειδή τηρήσαμε γενικά τους χρόνους, τα αποδέχομαι όλα. Το λόγο έχει για ένα λεπτό ο κύριος Πόλτσακ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο χαρακτήρας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι οικουμενικός και ο σεβασμός του το ίδιο. Μας προκαλεί αποτροπιασμό η περίπτωση του Ιμπραήμ Χαλάουα και οι συναφείς περιπτώσεις. Πρόκειται για έναν Ευρωπαίο επίκο που ταξίδεψε στο εξωτερικό και συνελήφθη άδικα και έχει υποστεί τέτοιες κακουχίες τα τελευταία δύο χρόνια. Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε διαβήματα προς τις Αιγυπτιακές αρχές. Αλλιώς ε, θα είναι δύσκολο οι πολίτες μας να ταξιδεύουν ε, στην Αίγυπτο όταν επικρατούν τέτοιες ε, συνθήκες. Δεν μπορώ να φανταστώ καν τη ζωή του ανθρώπου αυτού, ενός νεαρού που βρίσκεται στις φυλακές υπό άθλιες συνθήκες, περιμένοντας να δικαστεί. Δεν είναι η πρώτη περίπτωση δυστυχώς αυτή του Ιμπραήμ Χαλάουα, ούτε θα είναι η τελευταία. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για τέτοια καταστρατήγηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είχαμε και έναν πολίτη από βαλτικές χώρες που επίσης είχε ε, φυλακιστεί άδικα. Θα πρέπει να επισκεφτόμαστε τις φυλακές που πιο συχνά στην Αίγυπτο. Κύριο κύριος Μαριά. Πρόεδρε, συζητούμε για τον Ιρλανδό υπήκο Ιμπραήμ Χαλάουα, ένα πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αντιμετωπίζει δυνητικά τη θανατική ποινή στην Αίγυπτο για τη συμμετοχή του σε μια διαδήλωση στο Κάιρο οι αιγυπτιακές αρχές δεν έχουν προχωρήσει ακόμη στη δίκη του χαλάουα αφού αυτή αναβάλλεται συνεχώς ενώ υπάρχει πιθανότητα σε περίπτωση καταδίκης να του επιβληθεί η θανατική ποινή. παράλληλα η κράτησή του έχει διαρκέσει ήδη δύο χρόνια. καλούμε λοιπόν τις αιγυπτιακές αρχές να αφήσουν ελεύθερο τον ιμπραήμ χαλάουα και συμπαραστεκόμαστε στον αγώνα των συναδέλφων από την ιρλανδία επισημένοντας επιπλέον κύριε πρόεδρε ότι η ευρωπαϊκή ένωση πρέπει να επιδιώξει την κατάργηση της θανατικής ποινής όπου αυτή εφαρμόζεται και να ζητήσει από τις χώρες που την εφαρμόζουν ακόμη να συμμορφωθούν προς τα διεθνή πρότυπα. ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει για ένα λεπτό ο κύριος Γιάκοφτσιτς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο Ιμπραήμ Χαλάουα είναι Ιρλανδός υπήκος. Υπήκος δηλαδή μια χώρα μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και είναι υποχρέωση και καθήκον μας, πέραν αυτή τη συζήτηση που είναι απαραίτητη να γίνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να ζητήσουμε από την ύπατη εκπρόσωπο, αλλά και από την Επιτροπή μας για την Αντιπροσωπεία για Συνεργασία με την Αίγυπτο, αμέσως να θέσουν επιτάπητος ε, το θέμα αυτό στις Αιγυπτιακές Αρχές και να δούμε πώς θα αποφυλακιστεί το συντομότερο δυνατό και πώς θα εμποδίσουμε την, ε, την εφαρμογή της φρικτής απειλής της θανατικής καταδίκης. Θέλουμε την Αίγυπτο, θέλουμε την Αίγυπτο σε τέρο, θέλουμε να συνεργαστούμε μαζί μας, αλλά δεν έχει μόνο δικαιώματα η Αίγυπτος, έχει και υποχρεώσεις. Δεν μπορεί να φυλακίζει έτσι υπηκόους ε, ε, Ευρωπαίους. Θα πρέπει λοιπόν με διάταγμα το συντομότερο δυνατό να διαλευκάνει αυτή τη θέση. Θα είναι ε, η απόδειξη ότι θέλει να συνεργαστεί η Αίγυπτος με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το λόγο έχει για ένα λεπτό η κυρία Μαγκίνες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ακούσα τη ζήτηση αυτή και Ήθελα να πάρω το λόγο για να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο και την υποστήριξη από όλα τα κράτη-μέλη, από όλε τι πολιτικέ ομάδε για την ειλικρινή ανησυχία που εκφράζουν για ένα Ιρλανδό υπήκο. Υπήκο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελπίζω σήμερα να ενθαρρυνθεί η οικογένειά του από την σημερινή παρουσίαση και ελπίζω, και αυτό είναι πιο σημαντικό, να κατανοήσουν οι Αιγυπτιακέ αρχέ τι ανησυχίε μα. Θα πρέπει λοιπόν να τι ε, καλέσουμε να καταλήξουν ε, στην απόφαση να απελευθερώσουν τον κύριο Χλάβα. Γιατί όπως μιλάμε ε, σήμερα, αυτός βρίσκεται ακόμα στη φυλακή. Δεν μπορώ να φανταστώ πώς είναι η ζωή του. Χθες ε, στο Γραφείο Ζαχάροφ ακούσαμε μια παρόμοια υπόθεση. Ευχαριστώ λοιπόν το Κοινοβούλιο και ελπίζω να υπάρχει αντίκτυπος ε, της συζήτησης αυτής και να πετύχουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε. Το λόγο έχει για λεπτό η κυρία Thank you, Chair. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ελπίζω ότι η σημερινή συζήτηση θα δώσει κάποια ανακούφιση στην οικογένεια του Ιμπραχήμ, κάποια, κάποιοι των οποίων βρίσκονται εδώ σήμερα. Αλλά να σας υπενθυμίσω ότι πρόκειται για ένα θέμα όχι μόνο με τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά αυτό, αυτή η υπόθεση έχει να κάνει και με τα δικαιώματα του παιδιού. 17 ήταν ο Ιμπραχήμ όταν συνελεύθηκε και φυλακίστηκε. Πόσοι άλλοι βρίσκονται στη φυλακή στην ηλικία αυτή και πόσοι άλλοι έχουν χάσει τη ζωή τους σε τέτοιες ηλικίε. Φανταστείτε να είναι κανείς παιδί και να βρίσκεται σε τέτοιες συνθήκες. Αν ήταν το δικό μας το παιδί. Και ο Ιμπραχήμ είναι Ιρλανδός ε, υπήκος. Ελπίζω λοιπόν οι Αιγυπτιακές αρχές να εισακούσουν τις ανησυχίες μας και να λάβουν υπόψη ναι, τα όσα εκφράζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά να υπενθυμίσω ότι δεν πρόκειται μόνο για τα θεμελιώδη δικαιώματα ενός ενήλικα, αλλά και ενός παιδιού. Το λόγο έχει για ένα λεπτό η κυρία Κλούν. Σα ευχαριστώ και σα ευχαριστώ και την ευκαιρία που μου δίνετε να συμμετέχω στη συζήτηση αυτή. Να συμφωνήσω και με όλου όσοι υποστήριξαν την υπόθεση αυτή και να συγχαρώ την κυρία Μπόιλεν που μας ε, έθεσε το θέμα αυτή και να καλωσορίσω και την οικογένεια του Ιμπραχήμ ε, Χαλάβα που βρίσκεται εδώ σήμερα. Το πιο σημαντικό στοιχείο που αναφέρθηκε εδώ στη συζήτηση είναι ότι αυτός ο νεαρός ήταν ανήλικος, ήταν παιδί όταν συνελήφθησε και φυλακίστηκε και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να είναι το πρώτο μας επιχείρημα. Βρίσκεται στη φυλακή για μεγάλο χρονικό διάστημα, είναι πλέον 20 ετών και όπως και οι υπόλοιποι συνάδελφοι καλώ τις Αιγυπτιακές αρχές να αναγνωρίσουν ότι είναι Ιρλανδός και Ευρωπαίος πολίτης. Και να απελευθερέσουν τον Ιμπραχήμ να επιστρέψει στην Ιρλανδία και στην οικογένειά του κατανοώ το γεγονός ότι υπάρχουν και τα δικά τους συστήματα αλλά αυτή η διαρκής αναβολή της δίκης αποτελεί μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση και για το άτομο αυτό αλλά ήταν ανήλικος 17 χρονών είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το επιχείρημα Κύριε Επίτροπε Διαπιστώστε κι εσείς την ομοφωνία όχι μόνο των συναδέλφων από την Ιρλανδία αλλά όλων των περίγων του Κοινοβουλίου έχετε το λόγο να μας πείτε τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, Και εμείς ανησυχούμε πολύ για το ότι ενδεχομένως ένας δικός μας πολίτης αντιμετωπίζει τη θανατική ποινή. Πρόκειται για έναν Ιρλανδό και Αιγύπτιο πολίτη, ο οποίος εκτεί μακρά ποινή, αλλά ενδέχεται να καταδικαστεί και σε θάνατο. Παρακολουθούμε από την φυλάκιση του από το 2013 την κατάσταση του Ιμπραήμ Χαλάουα η ύπατη εκπρόσωπος, ε, η Φεντερίκα Μογκερίνη, παρακολουθεί την ε, περίπτωση του ε, στενά μαζί με τις Ιρλανδικές αρχές. Το θέμα το αντιμετωπίζουμε σε επίπεδο προξενικών αρχών και συνεργαζόμαστε πλήρως με την Ιρλανδία κατά συντονισμένο τρόπο. Προσπαθήσαμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα και ευρύτερα ως προς την αντιμετώπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αίγυπτο. Την, το προηγούμενο μήνα ξεκινήσαμε έναν διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα με την Αίγυπτο για πρώτη φορά μετά από πέντε χρόνια και θα θέλαμε η Αίγυπτος να ανταποκριθεί στα, στις διεθνείς προδιαγραφές για την αμεροληψία στις δίκες και θα πρέπει να υπάρχει ε, δίκαιη δίκη χωρίς ε, να επιβάλλονται μαζικές ποινές. Αντιτασσόμαστε στην θανατική ποινή για οποιοδήποτε λόγο και θα ασχοληθούμε με το θέμα της δικαιοσύνης στην Αίγυπτο μέσα στα πλαίσια της ε, συμφωνίας με την Αίγυπτο. Θα δούμε και το θέμα από πλευράς δικαιοδοσίας και στα πλαίσια της αντιμετώπισης των ανηλίκων και της επιβολής ποινή σε ανήλικο, τον οποίο αντιμετωπίζουμε ως ενήλικο. Ο Ιμπραχήμ Χαλάουα ήταν 17 χρονών όταν ε, συνελήφθη. Αντιτασσόμαστε στις μαζικές δίκες που παραβιάζουν το δίκαιο γιατί δεν λαμβάνουν υπόψη τις μεμονωμένες αξιόπινες πράξεις και καταφέρονται μαζικά κατά των κατηγορουμένων. Πιστεύω ότι αυτές οι μαζικές δίκες παραβιάζουν το άρθρο 9 της Διεθνούς Σύμβασης για τα ε, πολιτικά και αστικά δικαιώματα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για τη βελτίωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αίγυπτο και βασιζόμαστε στη συνεχή σας υποστήριξη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον ε, Επίτροπο Στυλιανίδη. Σας καλημερίζω και εγώ έχω λάβει 7 προτάσεις ψηφίσματος με την κατάληξη